Okay, Καλώς ορίσατε συνάδελφοι στο κοινό σκέλος της συνεδρίασης της ΑΦΕΤ και ΔΕΒΕ και την περασμένη εβδομάδα ή την προπερασμένη είχαμε κοινή συνεδρίαση για τις τροπολογίες της έκθεσης αυτής. Ε, Έχουμε δύο συνεισηγητέ για την αντιμετώπιση των μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών. Είναι η κυρία Βαλενσιάνο και ο κύριος Διευτεμέρα. Έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες. Θέλει κανείς από τους συγητές να πει τίποτα πριν αρχίσουμε να ψηφίζουμε και δεν σας βλέπω. Αγουστίν, που είσαι. Θες να πεις τίποτα πριν την ψηφοφορία ή να σοπάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Παρακαλώ, την προσοχή σας. Ε, μια και έχω το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελένα Βαλενθιάνο. Ήταν πολύ αποτελεσματική και επικοδομητική η συνεργασία μας. Ένα θέμα που στην αρχή ήταν δύσκολο και στη συνέχεια περίπλοκο ήρθε σε αίσιο πέρας εάν επικυρωθεί κατά τη διάρκεια της απογευματινής μας ψηφοφορίας και νομίζω ότι μπορούμε να ε, έχουμε ένα αποτέλεσμα μετά από εξυγερασμό συμφερόντων σε ένα τόσο περίπλοκο πρόβλημα. Και ε, επικεντρωθήκαμε στα ουσιαστικά και αφήσαμε στην άκρη τα επουσιώδη. Ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Υπάρχει προφορική τροπολογία, θα τη δούμε στο τέλος. Έτσι, αρχίζουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες μας. Πάμε. 108, all those in 108 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε. 127 ε, και 128 μαζί ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129 it 130 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Χρειάζεται επαλήθευση. 131 αρχίζει τώρα, παρακαλώ. Ωραία, να δούλευε και το μηχάνημά μου. Κάρτες βάλατε όλοι. Δεν βλέπω και πού είναι η καταμέτρηση. Α, πέρας. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά να το ελέγξουμε παρακαλώ. 134 αρχίζει ψηφοφορία. I Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Α, είναι πολύ μικρή διαφορά. Άξιζε να το ελέγξουμε. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε στην 152 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβεστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 167 υπέρ. Against. Abstentions. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά, αποχές. Έλεγχος, παρακαλώ, την 168. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι όσοι θέλατε πέρας. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 193 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα πάμε στη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.23 23 και 24 μαζί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 2.25 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.26 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 ε, υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τώρα έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα στη 241. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε στη 241. Πάμε. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ ε, αρχίσαμε. Ευχαριστώ. Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα της 241 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. 2.45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 251 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 272 και 273 μαζί υπέρ κατά Αποχές ε, εγκρίνεται. 2.74 επέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.75 επέ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 277 και 278 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.79 υπέρ κατά αποχές έλεγχος τη 279 ελέγχουμε αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 ειπε κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 292 μαζί με την 304 ταυτίζονται υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 296-297 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. η 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 302 και 299 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η 303 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Την 303 παρακαλώ επαληθεύουμε. Δεν κατάλαβα τι ψηφίζατε. Α, τώρα κατάλαβα. <laughs> Γιατί ε, Είχα αντιφατικά μηνύματα από εδώ. Ωραία, ζητώ συγγνώμη. Σοσιαλιστές δεν κατάλαβα τι έδειχναν υπέρ κατά. Συμβαστική 15 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα πάμε στην επόμενη σελίδα. Σε 3.32 κάτω κάτω υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 334 υπέρ. Τσεκ, ωραία. Ελέγχουμε την 333, αρχής ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Α, καταπίπτει. Ισοψηφία απορρίπτεται. απορρίπτεται. Ε, 334 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 3.34 αρχίζει τώρα. Has everybody voted? It was very close... Ψηφίσατε όλοι. Αν θέλετε να ψηφίσετε, ψηφίστε τώρα, γιατί έχουμε ισοψηφίε και μικρές διαφορές. Ορίστε. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 335 σε δύο τμήματα. Το τμήμα πρώτο, τη 335, αρχίζει ψηφοφορία. Όχι, ζητή συγγνώμη πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, τώρα για την 335, το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα, της 335 πάντων, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι 336 και 337 μαζί, ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 338 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 339 υπέρ, κατά αποχές. Για να την ελέγξουμε παρακαλώ την 339. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 3.41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα κερδίσαμε δύο σελίδες. Πάμε στην 3.62 και 3.63. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 364 σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ Against. Abstention. Κατά αποχές, εδώ χρειάζεται έλεγχος, το δεύτερο τμήμα του νέου Προέδρου. 364 είναι η τροπολογία. As everybody... Ψηφίσατε όλοι, παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 458 καταπίπτει. 366 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 384 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 388 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 406 in favor, against, 406 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 407 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4, 12 καταπίπτει, 408 υπέρ κατά αποχές. Κανείς δεν δείχνει τι ψηφίζεται, γι' αυτό θα τσεκάρω την 408. Παρακαλώ οι σοσιαλιστές να βλέπω πώς ψηφίζεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 409 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 410 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να το ελέγξουμε παρακαλώ αυτό. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Πάλι περσεύει ένα αυτό, το ΕΛΚ. Τι θα γίνει με την περίπτωσή σα. Α, τώρα εντάξει. Πέρα. Απορρίπτεται. Καλά, δεν σα χρειαζόταν ο έξτρα. Το δεύτερο τμήμα 4-10 υπέρ κατά. Το δεύτερο τμήμα της 4-10 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 422 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 423 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 424 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 425 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 428 υπέρ κατά πέκτη ζητώ συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.32 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 4.31 και 4.34 Πανομοιότυπες υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. 4.35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.36 υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. 4.37 υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.50 υπέρ, κατά, Εποχές. απορρίπτεται. Έλεγχος, εντάξει. Δεν κινήθηκε κανείς από αυτή την πλευρά, αλλά να ελέγξουμε για τα 450, έρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Δίκιο είχατε, αλλά πρέπει να σκόνετε τα χέρια. 451. Υπέρ ξεχωριστή, κατά τμήματα μάλλον ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4.53 και 4.54 ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.56 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 4.57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 4.59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4.60 και 4.61 επανομοιοτυπε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα. 4.60. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Α, δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε γιατί καλύπτεται τη συμβαστική. 462 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 463 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 464 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 465 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 466 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 467 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4,77 ε, και 4,87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4,78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4,79 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Έλεγχος για την 479. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 480. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 482. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 497. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος για την 497. Άρχεται η προφορία. Δεν ψήφισαν απαντές. Πέρας. Απορρίπτω. 4,98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4,99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 500 υπέρ κατά αποχέ. απορρίπτεται. 501 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 508 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 509 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5, 10, 5, 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 512 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 513, 514 ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. εγκρίνεται. 5.33 υπέρ, κατά απόχέ, απορρίπτεται. 5.34 υπέρ, κατά εποχέ Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε για την 534. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μεγάλη διαφορά. Ναι, Ελισλά, είναι στο λόγο. Διαδικαστικό. Ναι, με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Ναι, λίγο να μετακινηθώ ήθελα και στην κάμερα, διότι δεν φαινόμαστε και μετράνε ψήφι μας. Εγώ κοιτάζω πολύ προσεκτικά όμως κάθε σας κίνηση. Βλέπω ότι ψηφίζετε. Ο κάμεραμαν μπορεί να κάνει και αυτό που νομίζει. Συμβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5.40-481 πανομοιότητες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Εγκρίνονται. 541 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 542 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 543, 483 πανομοιότητες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 544, 484 πανομοιότητες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 545, 485 πανομοιότητες. Υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνονται. 546-486. νομιότυπε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 547. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Περνάμε σε θεολογικές σκέψει. Συμβαστή 29. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 και 42 πανομοιότυπες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνονται. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, απόχέ να ελέγξουμε. Ελέγχουμε για την 68, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. έγραφε. Απορρίπτεται. Δεν είχα δει καλά. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε για την 75. Άρχεται η πληροφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Έλα να ελέγξουμε για την 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύσκολο γιατί ήταν πολλές αποχές. Πέρας. Απορρίφθηκε. Οι εποχές έκαναν τη διαφορά. 77, 74 ε, εγκρίνονται. 36 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, κατά, συγγνώμη, αποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ετυλογικές αναφορές. Ετυλογικές αναφορές 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές ε, ε, Προφορική τροπολογία 2. Συνεισηγητές. Υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές Προφορική 3. Ε, υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. αποχέ, ε, απορρίπτεται. Οι γνωμοδοτήσει των επιτροπών τώρα τι είχα ξεχάσει. Και άλλε ψηφοφορίε. Γνωμοδότηση τη budget πρώτη. Παράγραφος 3 τη budget. Υπέρ, κατά, αποχέ, Εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχέ, Εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχέ, Εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, απόχέ, Εγκρίνεται. Η 7 καταπίπτει. Γνωμοδότηση Λίμπε. Παράγραφος 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία για την 18. Υπέρ. Κατά. Πρώτο τμήμα, με συγχωρείτε. 18. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έλεγχο. Έλεγχο για το δεύτερο τμήμα τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται.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 να ελέγξουμε, να ελέγξουμε για την 33 της ΛΥΜΠΕ, διότι έχετε κουραστεί και δεν βλέπω να σηκώνετε τα χέρια σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Όντω ήταν πολύ κοντά το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται με πολύ μικρή διαφορά. 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Και τώρα, συνάδελφοι, προφορική τροπολογία, νέα προφορική τροπολογία, η οποία υποβλήθηκε από τους συνεισηγητές. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βαλεντιάνου από τους συνεισηγητές. Ελένα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση ε, να λάβουμε υπόψη και τις τελευταίες αποφάσεις ε, της ε, διοίκησης Τραμπ. Λέμε λοιπόν, εκφράζει ιδιαίτερη, ιδιαίτερο προβληματισμό σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβερνήσεως των ΗΠΑ για πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου πολιτών από εννέα χώρες με πλειοψηφία, με μουσουλμανική πλειοψηφία ε, και την απαγόρευση λοιπόν να μπουν στην ε, χώρα. Ε, πιστεύει ότι τέτοιου είδους ε, ε, διαχωριστικές αποφάσεις δυναμητίζουν την κατάσταση σχετικά με την μετανάστευση και αυξάνουν την, τον ξενοφοβικό λόγο και οπωσδήποτε δεν συνάδουν με την Σύμβαση της Γενέβης. Θα πρέπει να ληφθούν οι υπόψη όλες οι, όλα τα συστήματα ε, διεθνούς προστασίας ε, και οτιδήποτε παρέχει νομική ασφάλεια. Και ζητούμε λοιπόν να υπερψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Θέλετε κύριε ε, Διάστα μέρα να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Συμφωνώ απολύτως. Άλλωστε πρόκειται για κείμενο επί του οποίου συμφωνήσαμε από κοινού. Υπέρ λοιπόν της τροπολογίας αυτής κατά αποχές ε, νομίζω ότι δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. everybody... Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ονομαστική, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με σοβαρή πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στους συνεισηγητές. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας στις συμβαστικές τροπολογίες που έκαναν αυτή την ε, ψηφοφορία συντομότερη από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Πολύ καλή συνεργασία μας. Ε, σας ευχαριστώ συνάδελφοι.